2015 για το Μαυροβούνιο. Εξ ονόματος του Συμβουλίου, το λόγο έχει η κυρία Χένης Φλασάρτ και Thank you again, Mr. President. Let me start by thanking you for the continuous and constructive contribution of the European Parliament to the advancement of Montenegro's accession process to the European Union and in particular your rapporteur Charles Tannock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 Ε, να ευθυγραμμίζεται με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουμε πλέον ανοίξει 22 από τα 35 κεφάλαια στις διαπραγματεύσεις. Σε ό,τι αφορά το μέλλον, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε μια ακόμα φορά την σημασία του κράτους δικαίου που είναι θεμελιώδης ε, αξία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και οριζόντια ενισχύα για όλη την ε, διαδικασία ένταξης. Όπως λέει και το ψήφισμα, η περαιτέρω πρόοδος θα συναρτηθεί από, από πρόοδος αυτό το θέμα. Το Συμβούλιο έχει δηλώσει ότι είναι πολύ σημαντικό όλο το κράτος δικαίου να δώσει συγκεκριμένα ε, αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος και της διαφθοράς. Χρειάζονται και άλλες προσπάθειες για να εστιάσουμε σε πραγματικές ε, μεταρρυθμίσεις με ρεαλιστικά αποτελέσματα μετρήσιμα. Το Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εξέλιξεις στενά. Σε ό,τι αφορά κάτι συναφές ε, συμμεριζόμαστε τον φόβο, ε, ε, την ε, επιθυμία μάλλον, το Μαυροβούνιο να συνεχίσει τις προσπάθειές του σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της κεντρικής διοίκησης και να ενισχύσει την ανεξαρτησία των θεσμών, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και την κατάσταση των, της ελευθερίας των μέσων μαζικής και ελευθερίας έκφρασης. Υπάρχουν και άλλες αδυναμίες, τις οποίες υπογραμμίζει και η Κομισιόν στην έκθεσή της. Ε, έχουμε κοινοβουλευτικές εκλογές αργότερα φέτος. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου της νέας εκλογικής νομοθεσίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το Μαυροβούνιο διέρχεται από μια δύσκολη, δυσχερή πολιτική κατάσταση και αυτό μπορεί να εμποδίσει τις μεταρρυθμιστικέ προσπάθειες. Είναι σημαντικό λοιπόν να επαναλάβουμε ε, ότι όλες, όλα τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να λάβουν τις ευθύνε τους και ε, να ξεκινήσουν ένα επικοδομητικό διάλογο ε, εντό του Κοινοβουλίου. Σε αυτό το πλαίσιο περιμένουμε ότι η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση θα συνεργαστούν ε, προκειμένου ε, να μην απογοητεύσουν ε, τις προσδοκίες του, του λαού. Αυτό άλλωστε είναι σημαντικό για να εξασφαλιστεί και η εμπιστοσύνη στην πολιτική διαδικασία και στο, στα όργανα του κράτους. Η επικοδομητική συνεργασία είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί η πολιτική δέσμευση που θα λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν που και που θα βοηθήσει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Ο διάλογος και η συμπερίληψη όλων ε, υπογραμμίζονται και στο ψήφισμα. Ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να περάσει αυτό το μήνυμα στο Μαυροπούνιο. Η σημαντική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, προκειμένου να ε, μέσω της ε, ε, ε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Εταιρικής Σχέσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να δούμε στο μέλλον και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η πρόοδος. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής έχει ο Επίτροπος κ. Χάν. Uh, Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Υπουργέ, αγαπητά μέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση για να συζητήσουμε για το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το Μαυροβούνι. Δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω ε, και τον εισηγητή για το Μαυροβούνι, τον κύριο Κίνοφ, για την ε, πολύ ισορροπημένη του έκθεση. Είναι ένα κείμενο το οποίο παρουσιάζει με τον καλύτερο τρόπο ε, την αξιολόγηση του 2015 για το Μαυροβίνι. Μαυροβούνι. Πριν από δύο χρόνια, αυτό τον Ιούνιο, θα έχουν ανοίξει οι ενταξιακές, προενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνι. Ήδη αναφέρθηκε από την Υπουργό ότι υπάρχουν 22 κεφάλια, κεφάλαια δύο ε, προσωρινά έχουν κλείσει. Όσον αφορά το κράτος δικαίου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, βρίσκεται στην ουσία, είναι η πεμπτουσία της διαδικασίας ε, ε, προσχώρησης τα τελευταία χρόνια υπήρξαν μεταρρυθμίσεις, εγκρίθηκαν νομοθετικές πράξεις και συστήθηκαν θεσμοί. Και όπως αναφέρθηκε επίσης ε, και όπως ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της του Νοεμβρίου, δεν τελειώνει εκεί η ιστορία. Η δική μας αξιολόγηση δυστυχώς λέει ότι η πραγματική μεταρρύθμιση σε θέματα κράτους δικαίου παραμένει περιορισμένη και αυτό αφορά την, τον αγώνα κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό το μήνυμα εκπέμπει ή εξέπεμπιζε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ποτκόριτσα. Όταν συναντώθηκα ε, με τον Πρωθυπουργό τον προηγούμενο μήνα, τον Συνεχάρη, για το ότι η χώρα του προσεχώρησε στο ΝΑΤΟ, <clears throat> επίσης είπα ότι η χώρα προχωράει και τώρα μπαίνουμε σε μια αποφασιστική φάση όσον αφορά στις ενταξιακέ διαπραγματεύσει και στο κράτο δικαίου. Πρέπει το Μαυροβούνι να σημειώσει αξιόπιστη πρόοδο στα κεφάλαια 23 και 24. Πρέπει να υπάρχει ε, χειροπιαστή το αρχείο μεταρρυθμίσεων και αυτό θα είναι όχι μόνο προς όφελος ε, των ε, διαπραγματεύσεων ε, προσχώρησης, να έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, διαφάνεια στη διοίκηση. Είναι ε, σαφές ότι πρέπει να καλύπτονται όλα τα κριτήρια που αφορούν στο κράτος δικαίου. Αυτά είναι τα προαπαιτούμενα για να προσελκύσει κανείς επενδύσεις για να δώσει όθηση στην ανάπτυξη. Όπως ξέρετε πολύ καλά, εγώ ε, προτιμώ να μιλάω για διαδικασία προσχώρησης και όχι διαπραγματεύσεις. Για τη τελική ανάλυση μιλάμε για την ε, οδό που ακολουθεί μια χώρα προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ένταξης. Ε, θα συνεργαζόμαστε με το Μαυροβούνι για να υπάρξει βελτίωση της ε, ανταγωνιστικότητάς του, να υπάρξουν τομεακές ε, μεταρρυθμίσεις, να βελτιωθεί η αγορά εργασίας όσον αφορά σε άλλα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων έχουμε δώσει οδηγίες στο Μαυρογούνι για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει ανοίγοντας ε, τα κριτήρια σύγκρισης, τα benchmarks. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να καλύπτονται από τη χώρα, κυρίως όταν μιλάμε για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο τόσο στην πολιτική ανταγωνισμού όσο και στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή. Όσον αφορά στην πολιτική κατάσταση στο Μαυροβούνιο, ο πολιτικός διάλογος που ξεκίνησε το Δεκέμβρη ε, ανεστάλλει χωρίς κάποια εξήγηση το Δεκέμβρη. Βέβαια, ε, παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί η συμφωνία ανάμεσα στους πολιτικούς ηγέτες σχετικά με τη σύσταση κυβέρνησης που θα χαίρει της εμπιστοσύνης του εκλογικού σώματος, είναι σημαντικό όλα αυτά σας λέω το ότι εξακολουθεί να υπάρχει κοινοβούλιο. Εφέτος στο Μαυροβούνι θα υπάρχουν γενικές και δημοτικές εκλογές. Ε, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί σωστά ο εκλογικός νόμος έτσι ώστε και οι εκλογές να είναι αδιάβλητες. Είναι λοιπόν ευθύνη των πολιτικών ηγετών του Μαυροβουνίου να διασφαλίσουν κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων πρώτος ομιλητής για την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Τάνοκ για τρία λεπτά. <clears throat> Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το 2016 θα είναι μια πολύ σημαντική χρονιά από πολιτική άποψη για το Μαυροβούνιο. Πλησιάζει στη δέκατη επέτειο τη ανεξαρτησία του και η χώρα αυτή όχι μόνο θα διοργανώσει βουλευτικέ εκλογέ, αλλά βρίσκεται και στη βορεία κρίσιμων διαπραγματεύσεων ε, ω προ την ένταξη στο ΝΑΤΟ μετά την πρόσκληση να προσχωρήσει στη Διατελετική Συμμαχία πέρυσι. Συνεχίζει λοιπόν την πρόοδό του. Έχουν ανοίξει 22 κεφάλαια και τα βασικά 23 και 24 και το 2016 θα ανοίξουν ε, καινούργια κεφάλαια και ελπίζουμε προσωρινά να κλείσουν ορισμένα από τα παλιά. Όπω αναφέρει και η έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ψήφισμά μα, η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα δημιουργούν σοβαρό προβληματισμό και ανησυχίε και κάποιε πτυχέ τη ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση. Πάντω υπάρχει γενική βελτίωση και πρόοδο. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη απαγγελία καταγγελιών για διαφθορά σε υψηλά κλιμάκια της διοίκηση και αρχίζει και λειτουργεί πλέον κανονικά το, ειδικό, το γραφείο του ειδικού εισαγγελέα. Και μάλιστα με την ίδρυση την πρώτη πρώτου του τρέχοντο έτου, του Οργανισμού της Πάταξης Διαφθοράς ενθαρρύνομαι από την ε, ενίσχυση του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Βέβαια, έχουμε κάποιε ανησυχίε ε, για τι διοικητικέ ικανότητε αυτών των θεσμικών οργάνων εξαιτία τη ελληπού χρηματοδότηση. Υπάρχουν οικονομικέ δυσκολίε και είναι φυσιολογικό μια μικρή χώρα σαν το Μαυροβούνιο να έχει τέτοια προβλήματα παρά την ε, ειδική ε, ενίσχυση και τεχνογνωσία που στέλνουν η Κροατία και η Σλοβενία. Πάντως ε, είναι προς τιμή του που το Μαυροβούνιο έχει γίνει υπόδειγμα σε ό,τι αφορά την ευθυγράμμιση της πολιτικής του με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωση και των κρατών μελών και έχει αποδείξει την ικανότητα σωστή συνεργασίας με τον γειτόνα τη στα θέματα αυτά. Επίσης, με μεγάλη γενναιότητα ευθυγραμμίστηκε πλήρως με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το κυρώσεων προς τη Ρωσία μετά την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας παρά τις, ε, τους στενούς δεσμούς που είχε με τη Ρωσία και συνεχίζει τη στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της διεθνούς διχατιστικής τρομοκρατίας. Ε, ε, ίσως γίνει του χρόνου δημοψήφισμα για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η θέση μου του είναι σαφής ότι είναι εσωτερικό ζήτημα του, Μοντε, του Μοντενέγρου, του Μαυροβουνίου και δεν είναι κάτι στο οποίο θα έπρεπε να επέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτου λεχθέντος θα πρέπει να έχουμε υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης και τις εξωτερικές επιρροές που θα ασκηθούν στο μικρό, στη μικρή αυτή τη χώρα, το Μαυροβούνιο. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ψήφισμα που εξετάζουμε και ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε επικοδομητικά με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες για να υπερψηφιστεί αυτή. Είναι η επιτυχής ιστορία των Δυτικών Βαλκανίων το Μαυροβούνιο. Μετά την πίεση όμως που άσκησε η προσφυγική κρίση σε όλα τα Βαλκάνια, το Μαυροβούνιο αρχίζει και αναδύεται όλο και περισσότερο ως φάρος σταθερότητας. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Ο κύριος Κόβατσεφ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μα, τον κύριο Τάνοκ, για την αγαστή συνεργασία που είχαμε. Πολύ συχνά αναφέρθηκε ότι το Μαυροβούνιο είναι ένα success story. Μία ε, επιτυχής ε, ιστορία. Βέβαια, δεν είναι αυτό κάτι δεδομένο. Θα πρέπει κάθε μέρα να γίνεται προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση και τη δημοκρατία. Η αντιπολίτευση ζητά τώρα διεξαγωγή νέων εκλογών. Και τίθεται να αμφιβόλω ακόμη και η ενταξιακή πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Φαίνεται ότι υπάρχουν τάσεις προς ανατολισμού προς τη Ρωσία. Παρ' όλα αυτά, η χώρα προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί με την κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Θα πρέπει να γίνει υπόδειγμα για χώρε όπω η Μακεδονία και η Σερβία για καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να στηρίξουμε την ενταξιακή πορεία και τον προσανατολισμό του Μαυροβουνίου για να συνεχίσει την πρόοδό του και να μην γίνουν οι κάτοικοι του θύματα των εξωτερικών πιέσεων από τρίτε χώρε. Ο κύριο Ανδρουλάκη, για δύο λεπτά. Το Μαυροβούνιο είναι ο Πρωταθλητή των Δυτικών Βαλκανίων στην πορεία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο γεγονό που επιβεβαιώνεται από το άνοιγμα 22 κεφαλαίων και το προσωρινό κλείσιμο 2. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζεται σε μια κρίσιμη στιγμή για το Μαυροβούνιο. Οι εκλογέ που θα διεξαχθούν μέσα στο τρέχον έτο είναι κρίσιμε για τη σταθερότητα και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν στο καλύτερο δυνατόν πολιτικό κλίμα. Η σοσιαλιστική ομάδα χαιρετίζει τι προσπάθειε τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια στην πορεία τη για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει όμω να αποφύγουμε τη μεταρρυθμιστική κόπωση η οποία μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια. για τον λόγο αυτό στο ψήφισμα εκτό των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει τονίζουμε την ανάγκη επιπλέον προσπαθειών στου τομεί τη δημόσια διοίκηση τη ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη τη καταπολέμηση τη διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματο. περιμένουμε ακόμα δράσει για την αντιμετώπιση τη φοροδιαφυγή των υψηλών κοινωνικών ανισοτήτων τη μακροχρόνια ανεργία και τη φτώχεια η κοινωνική πρόοδος για μας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας της ενταξιακής διαδικασίας. τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της ένταξης του μαυροβουνίου στο νάτο. δεν είμαστε αντίθετοι σε καμία περίπτωση στην ένταξή του στη συμμαχία όπως κάποιοι εδώ μέσα θέλουν να παρουσιάσουν. θεωρούμε όμως ότι είναι μια απόφαση που κάθε χώρα πρέπει να λαμβάνει μόνη της χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση. αυτό με το οποίο διαφωνούμε είναι η προσπάθεια σύνδεσης αυτών των δύο διαφορετικών διαδικασιών σήμερα εδώ συζητάμε για την ενταξιακή πορεία του μαυροβουνίου στην ευρωπαϊκή ένωση. ευρωπαϊκή ένωση και νατο είναι δύο διαφορετικοί οργανισμοί με διαφορετικούς στόχους. οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο υπονομεύει την αυτονομία του ευρωπαϊκού οράματος. για τον λόγο αυτό έχουμε καταθέσει μια τροπολογία που κάνει σαφή την παραπάνω θέση. Σα ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ κύριο Σεράντος για δύο λεπτά. Είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ για την πολύ αξιόλογη έκθεση που κάνει μια πλήρη επισκόπηση της κατάστασης στο Μαυροβούνιο και τον ευχαριστούμε γιατί δέχτηκε τη συμβολή μας ε, στην έκθεση αυτή. Το Μαυροβούνιο είναι η πιο προηγμένη χώρα στην ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι αν ευοδοθεί η διαδικασία της ένταξης του Μαυροβουνίου θα επηρεάσει θετικά και τις γειτονικές χώρες στην ίδια πορεία, δηλαδή και το Κωσυφοπέδιο και τη Βοσνία Αρζεγοβίνη. Βέβαια πολύ εύστοχα αναφέρονται στην έκθεση όλα τα εκρεμή ζητήματα και συμφωνώ με τον κύριο Χάν ότι βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή της ενταξιακής του πορείας στο Μαυροβούνιο και θα πρέπει να δείξει περισσότερες ε, ε, πρόοδους ε, στο θέμα της ε, ανεξαρτησίας της δικοσύνης, της πάταξης διαφθοράς, ε, της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα για το Μαυροβούνιο, πιστεύω, είναι οι εκλογές. Γιατί από την ανάκτηση της ανεξαρτησίας η χώρα αυτή ήταν βαθύτατα διχασμένη και πολλωμένη. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, γι' αυτό και οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι η πιο σημαντική και κρίσιμη πολιτική διαδικασία για τη χώρα αυτή. Όταν ε, διεξαχθούν διαφανείς ε, δίκαιες και ελεύθερες εκλογές, ε, τότε θα μπορέσουμε να πούμε ότι το Μαυροβούνιο θα έχει ένα δημοκρατικό μέλλον και η πορεία, η ενταξιακή του πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ πιο καθαρή. Είναι ευκαιρία αυτή για το Μαυροβούνιο να γίνει δημοκρατική χώρα και να επιτύχει στην ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ε, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυ και σε αυτή τη διαδικασία της προετοιμασίας και της διεξαγωγής ε, δίκαιων και σωστών εκλογών στο Μαυροβούνιο. Ο κύριος Κόουσο Περμουή για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, χαιρετίζουμε την πρόοδο του Μαυροβουνίου σε πολλούς τομείς. Πλην όμως ε, είμαστε επικριτικοί ακόμα ε, σε ό,τι αφορά τη σύνδεση μεταξύ της ένταξης των Ευρωπαϊκών και της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι δυνατόν ε, η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ να θεωρείται ότι ισχυροποιεί τη σταθερότητα στην περιοχή όπως αναφέρεται. Το αντίθετο. Πιστεύουμε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα στρατιωτικοποιήσει τα Δυτικά Βαλκάνια και θα δημιουργήσει περισσότερη αστάθεια. Καλούμε το Κοινοβούλιο να σκεφτεί το γεγονό ότι η κοινή γνώμη στο Μαυροβούνιο είναι διχασμένη σε ό,τι αφορά την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό λόγο θα πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα να αποφασίσουν. Αυτό είναι η δημοκρατία. Ω ομάδα διαφωνούμε επίση με τι πολιτικέ ιδιωτικοποιήσεων ε, οι οποίε προκαλούνται από την ενταξιακή διαδικασία. Τα οικονομικά αυτά μοντέλα έχουν αποδείξει ότι επιδρούν αρνητικά στους Ευρωπαίους πολίτες και συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη να επιβάλλονται σε κράτη τα οποία προσπαθούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας εμβαθύνουμε τη σχέση μας, ας στηρίξουμε την χώρα αυτή στι προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της. Ας ε, τη βοηθήσουμε να ενισχύσει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τον αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματο και της, ε, ε, και της διαφθοράς και στις προσπάθειές για την ελευθερία του τύπου και της έκφρασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Κυρίε και κύριοι, το Μαυροβούνι από μόνο του είναι μια πολύ πετυχημένη ιστορία. Δηλαδή είναι μια χώρα που εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεται σε διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σημειωθεί πρόοδο. Η έκθεση του κυρίου Τάνοκ, τον ευχαριστώ παρεπιπτόντω, είναι πολύ καλή, ισορροπημένη, αποδίδεται σημασία στον αγώνα ε, κατά τη ε, διαφθορά, του οργανωμένου εγκλήματο, τη ελευθερία του τύπου, τη ΜΚΟ. Περιλαμβάνονται όλα αυτά όπω και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ε, υπάρχει πρόοδο και στο θέμα των ΛΟΑ ΛΟΑΔ. Ε, όμως, όμως θα ήθελα να αναφερθώ περισσότερο στο, στα προβλήματα που υπάρχουν τώρα στο Μαυροβούνι. Υπάρχει μια πολιτική κρίση ε, και θέλω να επισημάνω ότι ένα αδελφό κόμμα δικό μας έχει καταθέσει μια πολύ επικοδομητική πρόταση για να διασφαλιστεί ότι όλα τα κόμματα θα συμπεριληφθούν σε μια μεταβατική κυβέρνηση, ότι θα βελτιωθεί ο εκλογικός νόμος για να επικρατήσουν δίκαιες και αδιάβλητες εκλογές. Ελπίζω αυτό το εγχείρημα να στεφτεί από επιτυχία γιατί είναι σημαντικό η διαδικασία να είναι τέτοια έτσι ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ότι η φωνή τους θα εισακουστεί. Σας ευχαριστώ πολύ και εμεί, ο κύριος Καστάλντο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Τάνο για τη δουλειά του σε αυτή την έκθεση όπου ε, πράγματι ε, έθεσε όλη του την εμπειρία για την έκθεση αυτή. Το Μαυροβούνι είναι ένα παράδειγμα στα Δυτικά Βαλκάνια από τις υποψήφιες χώρες. Αν δούμε λιγάκι το τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια θα δούμε ότι είναι η χώρα η οποία είναι πολύ πιο κοντά στο να προσεγγίσει την την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ένταξη. Πρέπει βέβαια να κάνει ακόμα πολλά όσον αφορά τη διαφθορά, ε, την δημόσια διοίκηση, τη λειτουργία της ε, που ε, εξακολουθεί να υπάρχουν εκεί προβλήματα. Δυστυχώς είναι κομματικοποιημένη και σχετίζεται άμεσα με τα κόμματα. Πρέπει να επισημάνουμε και το θέμα της υψηλής ανεργίας, κυρίως των νέων. Δυστυχώς δεν συμφωνώ εκεί που γίνεται λόγος για την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ, κυρίως όσον αφορά το χρονισμό. Κατά την άποψή μου ε, θα υπάρξουν εντάσεις με τις όμορες χώρες ε, και ε, ούμονον αυτό θα υπάρξει και πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας. Για να συνεχιστεί αυτός ο δρόμος πρέπει να υπάρχει συμφωνία, χρειαζόμαστε ένα μαυροβούνι δυνατό, δημοκρατικό που να μπορεί να κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις για να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο κύριος Σάπχαουζεν για 1,5 λεπτό. Η πολιτική σας για την ε, ε, διεύρυνση ε, θέτει σε σύγκρουση τη Δύση με την Ανατολή κάθε φορά. Κάθε φορά, χωρίς να λύσουμε τα παλιά προβλήματα, φεύγουμε προς τα μπροστά. Για παράδειγμα, ε, τα δίκτυα μετανάστευσης και το οργανωμένο έγκλημα στο Μαυροβούνιο, που είναι το επίκεντρο αυτών των δικτύων. Η, ε, η δυτική σας η δυτική πολιτική είναι μια ε, πολιτική που οδηγεί σε σύγκρουση με τον ευρωπαϊκό λαό και με την υπηρετική Ευρώπη. Η ρήξη έχει εγκατασταθεί σε μας ε, αντίθετα με την, ε, σε αντίθεση με αυτή την Ευρώπη το δημοψήφισμα της Δανίας, το δημοψήφισμα της Ολλανδίας για την Ουκρανία, ε, τα μελλοντικά το μελλοντικό δημοψήφισμα για το Brexit και αργότερα για την ε, Γαλλία, ε, πρέπει να δώσουν το λόγο στον, στους λαούς για να διαφωνήσουν με την κλεπτοκρατία του Μαυροβουνίου, με την αυταρχική Τουρκία κλπ. Και γι' αυτό το λόγο θέλουν να φύγουν οι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πια με Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δικτύων οργανωμένου εγκλήματος. Είναι η Ευρώπη την οποία ε, η Τουρκία καθιστά ε, ερήπιο. Την έχετε προδώσει την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Next speaker, Madam η κυρία Σούιτσα, για ένα λεπτό είναι η επόμενη ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ε, όταν μιλούμε για το Μαυροβούνιο, δεν μπορούμε παρά να γνωρίσουμε τη σημαντική πρόοδο που έκανε ω προ την και τη πορεία και σίγουρα θα πρέπει να στηρίξουμε ε, την πρόοδο της χώρας αυτής ε, στην προσπάθεια της ένταξης. Έχουμε σημαντική ευθυγράμμιση με την κοινή εξωτερική πολιτική και την κοινή πολιτική άμυνα. Βέβαια, πολύ δρόμο έχει ακόμη να διανύσει το Μαυροβούνιο για να φτάσει σε μια κατάσταση ε, πραγματικά πριν την ένταξη, παρόλο που έχει ξεκινήσει το, η διαπραγμάτευση τα 22 κεφάλαια. Εγώ κατέθεσα διάφορες τροπολογίες, μερικές τις δέχθηκε, άλλες όχι. Πάντως ευχαριστώ τον κύριο Τάνο για την πολύ αξιόλογη έκθεσή του. Θα ήθελα όμως ε, να τονίσω την ανάγκη ε, καλών ε, σχέσεων Μπορεί βέβαια με την Βοσνία Ριζεγοβίνη να, έχει, να έχουν αποκατασταθεί γειτονικέ σχέσει, αλλά εμεί έχουμε πρόβλημα διαφορά συνόρων με το Μαυροβούνιο που ε, παραμένει ακόμη εκρεμέ. Επίση, θα πρέπει ε, να αποζημιωθούν τα θύματα των ε, στρατοπέδων του Μαυροβουνίου. Είναι εκρεμές θέμα από τον Γιουκοσλαβικό πόλεμο. Επίσης, το θέμα του κόλπου του Κότορ ε, είναι μια ειδική διάρκεια περιοχή, το Μπόκα Θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη την πολυεθνωτική του ταυτότητα. Ας μην το ξεχάσουμε λοιπόν. Αυτά και ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να επισημάνω όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες. Ο κύριος Πίτσουλα, για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση του κυρίου Τάνοκ είναι ένα πολύ αξιόλογο και ισορροπημένο έγγραφο και ανέφερε τις ε, πρόοδους αφής που πραγματοποίησε πέρυσι το Μαυροβούνιο. Ε, εξακολουθεί όμως να υπάρχει ε, ένα υψηλό επίπεδο διαφθοράς που φαίνεται αντέχει στις μεταρρυθμίσεις. Έχουν ανοίξει 22 κεφάλαια, ακόμη και τα κεφάλαια 23 και 24 στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, πρόσφατα έγινε πρόσκληση από τον ΝΑΤΟ να προσχωρήσει το Μαυροβούνιο στην Διατλαντική Συμμαχία. Χαίρομαι γι' αυτό. Ε, γιατί θα έχουμε και εντό που φαίνεται ένα νέο μέλο στο ΝΑΤΟ. Πριν, ε, από 25 χρόνια έγινε επίθεση στην πατρίδα μου, στην ευρύτερη περιοχή τη Ιουκοσλαβία. Ε, είναι λοιπόν σημαντικό τα ανοιχτά θέματα να τα επιλύσουμε και με έναν νέο εταίρο. Έχουμε βέβαια το πρόβλημα τη οριοθέτηση των συνόρων, το θέμα τη κληρονομική διαδοχή από την πρώην Ιουκοσλαβία, η αποζημίωση των θυμάτων του πολέμου είναι μερικέ από τι εκκρεμότητε που υπάρχουν. Επίση, θα πρέπει να διαφυλαχθεί ο πολυεθνοτικό του κόλπου του Κότορ, τη περιοχή Μπόκα Κότορ είναι σημαντική και κρίσιμη αυτή η περίοδος για το Μαυροβούνιο. Θα πρέπει να επιλύσει πολλά εσωτερικά διλήμματα και αδιέξοδα και να χαράξει την ανταξιακή πορεία. Επίσης να έχει διάλογο με το, την κοινωνία των πολιτών για τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίο να πραγματοποιήσει. Σίγουρα σε αυτό ε, θα επηρεάσει και ε, το θέμα των σχέσεων κυβέρνηση και αντιπολίτευση, που δυστυχώ αυτή τη στιγμή είναι πολύ διαταραγμένε. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Τόμαση για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το Μαυροβούνιο βιώνει μια έντονη πολιτική κρίση και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή παρά είναι αισιόδοξο να αναμένουμε από τη χώρα αυτή πραγματική προσήλωση προς τις μεταρρυθμίσεις. Εμένα όμω ε, πρώτα απ' όλα με απασχολεί το γεγονός ότι δεν προσπαθεί αρκετά το Μαυροβούνιο να βελτιώσει τις σχέσεις ε, με τις γειτονικέ χώρες. Ε, η συνοριακή διαφορά με την Κροατία ούτε έχει καν αρχίσει να συζητείται. Παρ' όλα αυτά έχει ξεκινήσει τι έρευνε για υδρογονάθρακε και στην Αδριατική θάλασσα το Μαυροβούνιο, ε, συμπεριλαμβάνοντας 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τα κροατικά χωρικά ύδατα, παραβαίνοντας το πρωτόκολλο για το προσωρινό καθεστώς με τον νότια σύνορα του 2002. Το 2011 μάλιστα η Κροατία έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας για την παράβαση ε, της ε, προσωρινής χαρτογράφησης του πρωτοκόλου του 2002 στην προσπάθεια αξιοποίησης ε, των υδρογοναθράκων από πλευράς Μαυροβουνίου. Βέβαια η χώρα αυτή έχει δικαίωμα να εκμεταλλευτεί το φυσικό αέριο και, την, και το πετρέλαιο από την αντιρετική, αλλά φυσικά στα εσωτερικά χωρικά ύδατά του που δεν θα τα γνωρίσουμε αν δεν επιληθεί πρώτα η συνοριακή διαφορά. Ο κ. Κιουτσούκ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Χαν, κύριε Υπουργέ, συνάδελφοι. Το Μαυροβούνιο αποτελεί επιτυχημένη ιστορία σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις και την οικονομική σταθερότητα. Ε, και αυτό είναι πολύ θετικό για όλη την περιοχή. 22 κεφάλαια έχουν ανοίξει, συμπεριλαμβανομένων από των κεφαλαίων 23 και 24 για την δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις. Δύο κεφάλαια έχουν κλείσει προσωρινά. Το Μαυροβούνιο είναι επίσης παραδείγμα σταθερότητας και αξίζει το θαυμασμό μας. Η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια της χώρας ευθυγραμμίζονται με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήταν λογικό να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Όμως, έχει πρόσθετες ε, ευθύνες. Η κυβέρνηση θα πρέπει να βελτιώσει το κράτος, ε, συγγνώμη, το ρόλο του Εθνικού Κοινοβουλίου, να καταπολεμήσει την ε, διαφθορά και να εφαρμόσει τις κατάλληλες προδιαγραφές για την προστασία των μειονοτήτων και να εγγυηθεί τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή της χώρας. Κύριος Κάρβερ, για ένα λεπτό. Η συνεισφορά του Μαυροβουνίου στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη είναι σημαντική μας ε, ήδη από το παρελθόν μας ε, προστάτευσε από τον ε, πυρηνικό πόλεμο και το, συγγνώμη, το ΝΑΤΟ έχει συνεισφέρει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ε, όμως, πρέπει να επικρίνουμε και εκεί που χρειάζεται. Ε, δεν είμαι σίγουρος για την είσοδο του Μαυροβουνίου. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται σε μια πολύ ε, ε ανασφαλή περίοδο. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε καινούργιε συγκρούσεις. Ρεαλιστικά, τι μπορεί να συνεισφέρει ε, το Μαυροβούνιο στη συμμαχία από στρατιωτικής πλευράς. Ε, το ΝΑΤΟ είναι στρατιωτική συμμαχία και δεν είναι πολιτική ένωση. Ε, όμως ε, τα πολιτικά επιχειρήματα φαίνεται ότι είναι πιο ισχυρά από την πολιτική, ε, τη στρατιωτική λογική. Ευχαριστώ. Ο κ. Φερόν. Σεβόμαστε τον λαό του Ρουβουνίου που το 1892 ε, ε, κήρυξε τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λυπόμαστε όμως για την ε, απόφαση της χώρας να ε, χωριστεί από το σερβικό λαό. Σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή, πέραν των συνηθισμένων δηλώσεων, περιλαμβάνει και διάφορες αμφιβόλους ε, αξίας δηλώσεις σε ό,τι αφορά την αναγνώριση του κοσυφοπεδίου, την ε, απαγόρευση προνομιακών σχέσεων με τη Ρωσία, και την είσοδό του στο ΝΑΤΟ που είναι μια μηχανή που μασάει λαούς. Ε, το καταγγέλμα αυτό θα έχει πολύ αρνητικές συνέπειες. Ο κ. Μακάλιστερ, ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον Charles Στάνοκ. Το ψήφισμα του περιγράφει με ρεαλιστικό τρόπο την πορεία του Μαυροβουνίου προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου φαίνεται ότι πετυχαίνει. 22 ε, κεφάλαια από τα 35 έχουν ανοίξει και 2 έχουν κλείσει προσωρινά. Καλωσορίζω την απόφαση του ΝΑΤΟ να καλέσει το Μαυροβούνιο να ενταχθεί στην Βορειοατλαντική Συμμαχία η επιτυχία των διαπραγματεύσεων θα είναι, ελπίζω, το επόμενο βήμα. Σε ό,τι αφορά, επειδή είμαι για τη Σερβία, θα ήθελα να απογραμμίσω ότι 10 χρόνια μετά την ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου, οι δύο χώρε διατηρούν μια φιλική σχέση. Το πρωτόκολλο συνεργασία ε, για την ε, ε, σωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2015 και γίνονται τακτικά ε, επισκέψει ε, αξιωματούχων από τη μία χώρα στην άλλη. Ε, αυτό είναι, δείχνει πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα περιφερειακά προβλήματα των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κ. Μπετίνη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το ψήφισμα αυτό για το Μαυροβούνι κατά την άποψή μου είναι ισορροπημένο και είναι χρήσιμο για τον δρόμο που ακολουθεί αυτή η στρατηγική σημασία χώρα ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το Μοντενέγκρο, το Μαυροβούνι ζήτησε να μπει στο ΝΑΤΟ. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να αγνοήσουμε, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, ότι ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνοδεύεται και από τον δρόμο με το ΝΑΤΟ. Βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε για κοινωνική ένταξη. Το ΝΑΤΟ είναι στρατιωτικό συνασπισμό. Δεν μπορεί κανεί να χρησιμοποιεί την Ευρώπη για να έχει κατά νου το ΝΑΤΟ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και πρέπει να παραμείνουν έτσι. Αλλιώ θα είχε δίκιο η Ρωσία η οποία θα μπορούσε να καταγγείλει ε, τις ε, συμφωνίες μας ε, με τις όμορες προς εκείνη χώρα γιατί θα είχε δίκιο ότι πρόκειται για δούριους ύπους. Δεν έχουμε βέβαια το δικαίωμα να τα κανένα. Δεν πρέπει να κάνουμε τους ε, έξυπνους να επιδεικνύουμε χωρίς λόγο δύναμη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν μπορεί κανείς ε, να παραπλανήσει την Ευρώπη. Η Ρωσία είναι σημαντική για να αντιμετωπίσουμε και τον ISIS ε, και αν θέλετε και από διπλωματικής και τακτικής πλευράς. Ως εκ τούτου νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρθηκαν σήμερα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κούκαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ε, χάρη στον κύριο Τάνοκ έχουμε μπροστά μας μια πάρα πολύ καλή έκθεση και χαίρομαι που εστιάζεται σε προτεραιότητες όπως είναι η δικαστική εξουσία, ο γόνας κατά της διαφθοράς αλλά επίσης και σε άλλα κρίσιμα θέματα όπως είναι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη χώρα αυτή. Το Μαυροβούν έχει προχωρήσει στην προενταξιακή διαδικασία και πρέπει να το στηρίξουμε. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό αυτή την πρόοδο και εμεί. να τη χαιρετήσουμε κλείνοντας κάποια κεφάλαια που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Την ε, προενταξική διαδικασία του Μαυροβουνίου πρέπει να την δούμε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ε, Ας μην ξεχνάμε ότι έχει εναρμονιστεί πλήρως με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και άλλες χώρες της περιοχής, το Μαυροβούνι χαρακτηρίζεται από εσωτερικές πολιτικές διαμάχες ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι οι μάχες αυτές δίνονται στο κοινοβούλιο και αποκηρύσει κανείς τη βία στους δρόμους. Η κυρία Τζεντήλε για ένα λεπτό. Κοιτάξτε, υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη όσον αφορά τη συμφωνία με το Μαυροβούνι. Είναι απαραίτητο να καταβληθούν προσπάθειες για να μπορούμε να διασφαλίσουμε την ελεύθερη ε, συμμετοχή στις επόμενες εκλογές. Ε, να αποδίδεται σημασία στο ότι είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν πλήρως ε, τα δικαιώματα αλλά και η προστασία των εργαζομένων. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει ασφάλεια στο χώρο εργασίας, κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους εργαζόμενους. Θα ήθελα να πω ότι ανησυχώ λιγάκι ε, για το ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει απαραίτητη προστασία για τις μειονότητες και τις πολιτικές και τις εθνοτικές και την ε, ομάδα των ΛΟΑΔ. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη να προαχθούν τα δικαιώματα συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή, στη θεσμική ζωή αλλά και στην αγορά εργασίας. Ο κύριο Πλένκοβιτς είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τάνοκ για την κατάρτιση της έκθεσης. Σίγουρα το Μαυροβούνιο έχει προχωρήσει περισσότερο από όλες οι υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην ενταξιακή πορεία και μάλιστα έχουν ανοίξει προσωρινά μερικά κεφάλαια, ενώ άλλα έχουν ήδη προσωρινά κλείσει. Θα πρέπει φυσικά να συνεχιστούν οι συστημικές μεταρρυθμίσεις ε, ε, που άπτουν το κεφαλαίο 23 και 24, δηλαδή ε, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου. Μετά την σοβαρή πολιτική κρίση για την οποία γίναμε μάρτυρες στους τελευταίους μήνες, θα πρέπει να βρεθεί διακομματική συνένεση για την πρόοδο. Αυτό θα είναι σημαντικό στοιχείο της σταθερότητας αλλά και της κουλτούρας του διαλόγου στο Μαυροβούνιο. Επίσης, το θέμα της ένταξης στο ΝΑΤΟ θα συμβάλλει να σταθεροποιηθεί και το Μαυροβούνιο αλλά και η περιοχή της Αντιρρετικής γενικότερα. Επίσης το θέμα των μειονοτήτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και της ε, Κροατικής, ε, το θέμα της κληρονομικής διαδοχής από την πρώην η δίωξη των εγκληματιών του πολέμου ε, και οι πολυθνοτικός χαρακτήρες του κόλπου του Κότορ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Νίνα ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, το Μαυροβούνιο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώ ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προωθήσει θετικέ μεταρρυθμίσει σε μια τρίτη χώρα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το συλλογικό τη βάρο για να προωθήσει τη σταθερότητα, την ευημερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ευρύτερη περιοχή, κάτι που είναι προ το, ε, το συμφέρον όλων μα. Ε, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να το κάνει μόνο μία χώρα. Η στενή συνεργασία με το Μαυροβούνιο δεν έχει μόνο ε, θεμελιώδη χαρακτήρα λόγω της ε, συμμετοχής της χώρας αυτής στη Βαλκανική Οδό. Αλλά η χώρα αυτή μπορεί να είναι και κόμπος ε, λαθρεμπορίου όπλων που μπορεί να καταλήξουν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, έχουμε το ε, σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πάταξη του λαθρεπορείου όπλων που υιοθετήθηκε μετά τις επιθέσεις των Παρισίων. Χαίρομαι που πρόσφατα ε, άνοιξαν δύο διαπραγματευτικά κεφάλαια για τις μεταφορές και την ενέργεια και δίνουμε μια νέα όθηση στις σχέσεις μας με τη σημαντική αυτή για τον χώρα. Θα πρέπει φυσικά να συντελεστεί πλέον πρόοδος στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, του δικαστικού συστήματος και στην πάταξη της διαφθοράς. Και οι φετινέ εκλογέ θα είναι μια λιδία λίθο. Θα πρέπει να είναι δίκαιε και ελεύθερε ε, και να εξασφαλιστεί επίση η ανεξαρτησία και η ελευθερία έκφραση των μέσων μαζική ενημέρωση. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, Κύριο Πέτερλε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας, τον Charles Στάνοκ, για μία ακόμη καλή και αξιόλογη έκθεση με θέμα το Μαυροβούνιο, το οποίο συγχαίρω για το άνοιγμα νέων διαπραγματευτικών κεφαλαίων. Με το άνοιγμα νέων κεφαλαίων για διαπραγμάτευση θα συμβάλλουμε στην προώθηση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για να έχουμε ένα εύρυθμο κράτος δικαίου στην χώρα αυτή. Είναι σημαντικό να μην αναχαιτιστεί η ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου από την εσωτερική πολιτική κρίση και πόλωση. Θα πρέπει να αποκατασταθεί η πολιτική σταθερότητα της χώρας για να μην αναχαιτιστεί η ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Κριστέα. Συγχαρητήρια στον κύριο Τάνοκ για την ουσία της έκθεσης. Ακούγοντας την, τη συζήτηση και διαβάζοντας την έκθεση, βλέπουμε ξεκάθαρα που βρίσκεται το Μαυροβούνιο σε ό,τι αφορά την ένταξή του. Χρειάζονται προσπάθειες σε διάφορους τομείς, είναι σαφές. Για παράδειγμα, ε, διαφάνεια και λογοδοσία στη δημοσία διοίκηση, ανεξαρτησία στην ε, δικαιοσύνη, αξιόπιστη τη καταπολέμηση τη διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματο. Όμω από την αρχή των διαπραγματεύσεων το Μαυροβούνιο έχει διανύσει μεγάλο, μεγάλη απόσταση. 22 κεφάλαια άνοιξαν, δύο έχουν κλείσει προσωρινά. Είναι προφανώ στην ε, κορυφή του καταλόγου των, χωρών, των προσένταξη χωρών και η συνεισφορά του ξεπερνά τα σύνορά του. Αποδεικνύει ότι η, διαδικασία, η ενταξιακή διαδικασία είναι προβλέψιμη, είναι ακόμα αξιόπιστη. Ευχαριστώ. Thank you. And now we start the catch the eye procedure. Ξεκινάμε τη διαδικασία Catch the Eye. Ο κ. Πόσπιλ. Mr. Pospíšil. Pospíšil. Děkuji pěkně, ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή. Ε, μελέτησα ιδιαίτερα το θέμα της δικαιοσύνης και της καταπολέμησης διαφθοράς γιατί με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι αυτό εδώ και 10 χρόνια. Ε, ήταν, είναι σημαντική προσπάθεια που έχει γίνει και που πρέπει να γίνει. Δεντολογικός κώδικας για τους δικαστές για παράδειγμα είναι ε, σημαντική προϋπόθεση, όμως δεν πρέπει να μείνει στα χαρτιά, πρέπει πραγματικά να εφαρμοστεί. Θα ήθελε η Κομισιό να βοηθήσει όσο μπορεί το Μαυροβούνιο. Η Τσεχική Δημοκρατία ε, χαίρεται όταν ε, βλέπει δικαστές από άλλα κράτη να μας επισκέπτονται και να ε, ενημερώνονται για το πώς έχουμε μεταρρυθμίσει το δικό μας σύστημα και ας βοηθήσουμε λοιπόν το Μαυροβούνιο, μην σταθούμε μόνο στα λόγια, ας τα κάνουμε πράξη για να ενισχύσουμε το κράτος δικαίου εκεί. Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Επίτροπο ότι η διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ξεπερνά το, απλό, το στενό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Προϋποθέτει ανοιχτή αγορά, κοινέ πολιτικές, ε, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση και το καθεξής. Χαίρομαι που ε, μιλήσαμε για τα θέματα αυτά στη συζήτηση και κυρίως στην ανάγκη ε, μεταρρύθμισης και ανασυγκρότησης του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης. Ε, σημαντικό το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24, αν και είναι μάλλον μικρή η πρόοδος μέχρι στιγμής. Πάντως δείχνει την ετοιμότητα του Μαυροβουνίου να έχει διαφανή διαχείριση των οικονομικών του θα πρέπει να βοηθήσουμε το Μαυροβούνιο σε όλες τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές που θα χρειαστεί να κάνει. Επίσης, στην ενταξιακή πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λύσουμε τις εκκρεμότητες και τα ανοιχτά ζητήματα με τις γειτονικέ χώρες. Και για την Κροατία είναι πολύ σημαντικό το θέμα των συνόρων, της κληρονομικής διαδοχής από την πρώην Ιουκοσλαβία και η αποζημίωση των θυμάτων των στρατοπέδων του Μαυροβουνίου. Ευχαριστώ. Το Μαυροβούνιο, από ό,τι φαίνεται και από την έκθεση, έχει προχωρήσει πάρα πολύ στην ε, ενταξιακή του πορεία παρόλε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στον εκδημοκρατισμό του. Έχει αρχίσει και ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι, έχει, έχει αξία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει για να δώσει κίνητρο και σε άλλες γειτονικέ χώρες. προκειμένου ε, να ενδυναμώσει και να αναθερμάνει τις ενταξιακές διαδικασίες ε, των γειτονικών χωρών. Θα πρέπει να στηρίξουμε το Μαυροβούνιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Γιάκοβτσικ. Κύριε Πρόεδρε, το Μαυροβούνιο είναι ε, θαυμάσιο και χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει πώς ε, χάρη σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις επιταχύνεται ο εκδημοκρατισμός, ε, επιταχύνονται οι μεταρρυθμίσεις και μια χώρα προσαρμόζεται και ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και είναι παράδειγμα προς και για τις γειτονικές χώρες του Μαυροβουνίου. Την Αλβανία για παράδειγμα, που με τίποτα δεν ξεκινά τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη. Ελπίζω τέτοια θετικά αποτελέσματα να δούμε και στην Αλβανία και στη Βοσνία και Ριζεγοβίνη και στη Μακεδονία, λέει ο εισηγητής. Επίσης ήθελα να απευθύνω έκκληση και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση του Μαυροβουνίου, αυτή της φίλης χώρας. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω έκκληση προς τις δυνάμεις ε, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ε, για ειλικρινή διάλογο ε, θα πρέπει όλες οι πολιτικές παρατάξεις να συνεργαστούν για να διεξαγάγουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές για να επιταχυνθεί η ενταξιακή διαδικασία και η προσέγγιση του Μαυροβουνίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Πόλτσακ. Στην, στο προηγούμενο θέμα της ε, ήμασταν πολύ διστακτική σε ό,τι αφορά την ένταξή της. Σε αυτή την περίπτωση του Μαυροβουνίου θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την πρόοδο που έχει κάνει βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου των προσένταξη χωρών. Θα πρέπει να το συγχαρούμε. Ο κ. Πόσπισελ αναφέρθηκε στο θέμα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να μιλήσω για την αποπολιτικοποίηση και αποκομματικοποίηση της ε, δημόσιας διοίκησης. ο κρατικός μηχανισμός ε, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος ε, ε, πολιτικών παρεμβάσεων. Το Μαυροβούνιο θα πρέπει να βελτιώσει την κατάσταση. Ε, παρόλα τα πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που είναι πολύ κοντά στην ένταξη. Ευχαριστώ. Ο Σόλτερς. Ευχαριστώ. Το Μαυροβούνιο είναι παράδειγμα προόδου και επιτυχημένων προσπαθειών μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Όλοι επιθυμούμε να συνεχίσει με τον ίδιο ενθουσιασμό προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει βέβαια να υπογραμμίσουμε το θέμα της ε, καταπολέμησης της ε, διαφθοράς ε, και την ανάγκη να βελτιωθεί η κατάσταση στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, καθώς επίσης και στην διαδικασία εκδημοκρατισμού. Είναι μια εξαίρετη χώρα, η φύση είναι εκπληκτική, τη γνωρίζω πολύ καλά και ως Ευρωβουλευτής θα ήθελα να καλέσω όλες τις κρατικές αρχές και όλους τους πολιτικούς να μην ξεχνούν τους ε, φυσικούς θησαυρού και να τους προστατεύουν έναντι οποιονδήποτε αρνητικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ο λόγος στον Επίτροπο κύριο Χάν. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητά μέλη. Θα ήθελα να επαναλάβω στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως τον εισηγητή που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθάει το Μαυροβούνι να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το ψήφισμά σας αναφέρει τα σημαντικότερα στοιχεία ε, που αφορούν στην πολιτική της χώρας, έχουν γίνει πάρα πολλά, υπάρχουν όμως και προκλήσεις για το μέλλον. Το να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα της ε, χώρας ε, και τη στηρίζουν όλα τα κόμματα. Το Μαυροβούνι αυτή τη στιγμή ακολουθεί αυτό το στόχο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καθοριστική σημασία η δική σας υποστήριξη ε, για να υπάρξει διεύρυνση. Το Μάιο το Μαυροβούνι θα εορτάσει τη δέκατη επέτειο της ανεξαρτησίας του. Τα τελευταία δέκα χρόνια πέτυχε πάρα πολλά. Ξεκίνησε προενδιαξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δέχτηκε ε, πρόσκληση να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ. Επιτεύγματα αυτά. Αλλά όπως ήδη αναφέρθηκε από αρκετούς ομιλητές ε, εξακολουθούν να ε, μένουν αρκετές προκλήσεις. Δηλαδή η πλήρης εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ο οποίος θα διασφαλίσει ε, για το 2016 αδιάβλητες ε, βουλευτικές και δημοτικές εκλογές. Επίσης, ε, να επικρατήσει κράτος δικαίου, να υπάρξουν οικονομικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα από πολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Όπως ανέφερα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, το 2016 θα είναι το έτος χειροπιαστών αποτελεσμάτων κυρίως για θέματα κράτους δικαίου προσβλέπουμε στο να επιτύχει το Μαυροβούνι συγκεκριμένα αποτελέσματα ε, και χαιρόμαστε που το Κοινοβούλιο θα βοηθήσει το Μαυροβούνι για να επιτύχει το στόχο του. Ε, και εμείς ε, τώρα λοιπόν θα ήθελα να τον δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Όπως πολλοί από σας σημειώσατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υπάρχει μια θετική προοπτική του Μαυροβουνίου. Τώρα, το Μαυρούμι βέβαια έχει και πολλά ακόμα να κάνει, για παράδειγμα στο θέμα του κράτους δικαίου. Οι θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ιδιαίτερα οι δημοκρατικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κάνουν μοναδική και είμαστε περήφανοι για αυτές. Είναι σημαντικό λοιπόν το Μαυροβούνιο να προσαρμόσει το κράτος δικαίου του ε, με τρόπο πολύ συγκεκριμένο για παράδειγμα σε θέματα καταπολέμησης διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος. Πολλοί από εσά σχολιάσατε επίση το ΝΑΤΟ και τη σχέση του Μαυροβουνίου με το ΝΑΤΟ. Θεωρώ ότι το Μαυροβούνιο είναι φίλη χώρα που συνεισφέρει με πολλούς ε, τρόπους στην ε, εδραίωση ειρηνικών και φιλικών σχέσεων διεθνώς. Ε, ο ρόλος επίσης του Μαυροβουνίου στην γειτονία του είναι πολύ σημαντικός. Άρα η ένταξη του ε, άρα ο ρόλος του, του περιφερειακά είναι πολύ θετικός. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου, ε, που δεν είναι. Τώρα, στην πορεία προς την ένταξη, θα ήθελα να σας βεβαιώσω ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ στενά την πρόοδο του Μαυροβουνίου με ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα του κράτους δικαίου και σε άλλα σημαντικά ζητήματα που αναφέρονται και αναφέρθηκαν σήμερα και στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ.